ο κύριος Πρόεδρος. That was beautiful. Thank you so much. Mr. Combenet, you have to repeat this now. <laughs> no, in the original. Λοιπόν, θα πρέπει να το ξαναεπαναλάβετε εις ε, την ε, γλώσσα. Ε, τα συνοπτικά πρακτικά της θεσμής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Καλώς. Τότε τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΥΠΑ ε, της Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και τον αποκλεισμό της Γάζας. Θα ήθελα να παρακαλέσω την ε, είπατε εκπρόσωπο την κυρία Άστον να λάβει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι πολύ σοβαρή η συζήτηση της Γάζα, διότι συζητήσαμε ήδη το θέμα ή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Δευτέρας ε, και είμαι σε συνεχή επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν διάφορα ψηφίσματα. Θέλω λοιπόν να σας πω τι έγινε εκτός της Γάζας διότι είναι ε, απαράδεκτο και το λέω σαφώς. Ε, νέα άτομα ε, πέθαναν σε διεθνή ύδατα και πρέπει να υπάρξει μία έρευνα την οποία οι Ισραηλινοί, οι Παλαιστίνοι και οι Τούρκοι απαιτούν και καταρτίστηκε μία ανεξάρτητη επιτροπή με ε, δύο ανεξάρτητα ε, αλλοδαπά μέλη για να παρακολουθήσουμε ε, το, την πορεία προς τα πορίσματα και να αποφασίσουμε θα, σου, θα σας πω ότι η απώλεια ζωής ήταν τραγική. Πρέπει όμως να θυμηθούμε γιατί πήγαινε ο Στολίσκος στη Γάζα καταρχήν ε, και ε, ε, πάλι η Γάζα επανήλθε τώρα εις το επίκεντρο της συζητήσεως είναι το, πήγα ε, στην Γάζα πρόσφατα και αυτό που είδαμε σόκαρε διότι ε, δεν υπάρχει ούτε το εξαιρετικό εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει στο Ισραήλ ούτε καν η βασική εκπαίδευση. Χρειάζεται ε, το ΟΗΕ ε, υλικά για να μπορέσει να χτίσει οικισμούς, ε, σχολεία, νοσοκομεία και υγειονομικές υπηρεσίες ε, δεν ε, υπάρχουν ε, νοπά τρόφιμα και δεν μπορεί να υπάρξει ανοικοδόμηση και ο αποκλεισμός αυτός δεν είναι αποτελεσματικός και είναι λανθασμένος διότι πολλοί διέρχονται από παράνομα τούνελ το μπλοκάρισμα αυτό δίνει στη χαμά τη δυνατότητα να προσελκύσει την προσοχή. Και τέλος, η κατάσταση της Γάζα δεν καθιστά πιο ασφαλώς το Ισραήλ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Γάζα και να υπάρχει ασφάλεια για το λαό του Ισραήλ. Πρέπει δύο αυτές απαντήσεις να πάνε από κοινού, διότι αν τις διαχωρίσουμε θα αποτύχουμε Αποφασίσαμε λοιπόν ότι πρέπει να λάβουμε αυτή την πρωτοβουλία, να λάβουμε στεναρά μέτρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν θα είναι εύκολο να αρθεί ε, ο αποκλεισμό, διότι χρειάζεται τη συνεργασία πολλών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά εδώ και πολύ καιρό να υπάρξει άρση του αποκλεισμού αλλά τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Πρώτα πρέπει να ανοίξουν οι διελεύσεις για να μπορέσουν το ανθρωπιστικό προσωπικό και ε, οι πολίτες να ε, διακινηθούν ελεύθερα και το πιο βασικό χρειάζεται η συμφωνία του 2005 που συμφωνήθηκε μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και του Ισραήλ να ισχύσει διότι αυτό είναι το βασικό πλαίσιο ε, επιπλέον ε, υπάρχει μία ε, σύντομη λίστα απαγορευμένων υλικών τα οποία δικαιολογημένα το Ισραήλ να αρνείται να κυκλοφορήσουν και ελπίζω ότι με αυτό έχουμε κάνει ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Επίσης υπάρχει μία αποστολή στην Ράφα που θα μπορούσε να αναβιώσει και θα πρέπει να επανεστιάσουμε την αποστολή μας ή να δημιουργήσουμε μία άλλη. Θα δημιουργηθεί μία task force η οποία θα έχει την αναγκαία εμπειρία. Θα στείλουμε μία διερευνητική αποστολή σύντομα για να δούμε πώς μπορούμε με τον καλύτερο τρόπο να συμβάλλουμε σε μία λύση και υπέρ του λαού της Γάζα και καλύπτοντας τα συμφέροντα του Ισραήλ. Θα πρέπει να αποβλέπουμε στην ειρήνη διότι η Γάζα θα είναι ένα άρρηκτο Μέρο μέρος του μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους οπότε η Γάζα θα πρέπει να ε, προχωρήσει όπως προχώρησε η συμφιλίωση με τον Παλαιστινιακό λαό και αυτά είναι τα δύο θέματα που παραμένουν οι στόχοι μας και τέλος ε, εφόσον έχουμε ε, διατηρήσει τις συζητήσεις θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους Άραβες ομολόγους μας οι οποίοι συμβάλλουν και θα πρέπει να, να συγχαρούμε όλους οι οποίοι εργάζονται για την ειρήνη στην περιοχή και είμαι βέβαιη ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα με συνδράβει σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Των πολιτικών ομάδων ε, εκ ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Κασουλίδης για 1,5 λεπτό. Thank you, President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εάν κάποιος ε, θα έπρεπε να επιμείνει για την ανάγκη αμεριληψίας, ε, αξιοπιστίας και διαφάνειας ε, υπό τη διεθνή εποπτεία, αυτό θα έπρεπε να είναι το Ισραήλ. Ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Πράγματι το αποφάσισαν οι Ισραηλοί, αλλά χρειάζονται περισσότερα για να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη τη διεθνού κοινότητα. Ο αποκλεισμό τη Γάζας πρέπει να έρθει. Το δήλωσε και ο πρόεδρος Ομπάμα. Είπε ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη. Η Χαμάς είναι η μόνη ευνοούμενη από αυτόν τον αποκλεισμό. Χρηματοδοτείται, αυτοχρηματοδοτείται από τις ε, επικερδείς συναλλαγές, λαθρεμπορίου, μέσω διαφόρων ε, διάβλων και κυκλωμάτων που τελικά ε, διανέμει σε όσους Παλαιστινίους ζητούν αυτά τα αγαθά. Τελικά ε, τίποτα δεν έχουν ε, ε, κερδίσει. Ο Τζιλάτ Χαλίδ ακόμη στην φυλακή. Οι Ισραηλινοί δηλαδή έχουν κερδίσει. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε τους διεθνούς παράγοντες που προσπαθούν να διανοίξουν κάποιοι οδικοί διάδρομοι για την μεταφορά των ε, εμπορευμάτων και των αγαθών. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που τελικά θα οδηγήσει και στην ανοικοδόμηση της περιοχής. Στο μεταξύ προσπάθειες για τη συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων ε, παλαιστινιακών ε, ομάδων και φρατριών θα πρέπει να γίνουν. Οι ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια επίσης βέβαια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Keyser για δύο λεπτά. Δεν απευθύνομαι σήμερα σε εσά κύριε Πρόεδρε, ούτε σε εσά κυρία Άσον και σε ζητώ συγγνώμη. Σήμερα απευθύνομαι σε αυτούς που μα ακούνε, δηλαδή τα μέλη της, του στολίσκου του Μαρμαρά που είναι σήμερα εδώ. Σα απογοητεύσαμε και δεν σα ικανοποιήσαμε. Βλέπω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή μα τηλεφωνούσατε, ελπίζατε ότι ότι η Ευρώπη θα σας ε, προστάτευε αλλά η Σμάτιν μείνατε μόνοι χωρίς ε, όπλα ε, αντιμέτωποι με στρατιωτικούς οι οποίοι είχαν εντολή να ανοίξουν πυρ και μας ζητάτε σήμερα δικαιοσύνη διεθνή ανεξάρτητη δεν έχετε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη του Ισραήλ ακόμη και αν πλαισιώνονται από διεθνείς γιατί οι φίλοι σας ε, σκοτωθήκαν, ε, κατεστράφησαν ε, οι υπολογιστέ σας, οι φωτογραφικές σας μηχανές, τα φιλμ σας για να παρουσιαστεί η εικόνα που ήθελε να προβάλλει το Ισραήλ τρεις μέρες μετά και σας μεταχειρίστηκε σαν τρομοκράτες το Ισραήλ πολλές φορές σας σκότωσε και δεν καταλάβατε τι χρειαζόταν γινόταν. Ε, θα χρειάζεστε λοιπόν να υπάρχει δικαιοσύνη και να μπορείτε να πιστέψετε. Γι' αυτό και ορισμένοι από εσά σκοτωθήκαν και θέλετε άμεσα η πολιορκία της Γάζας να αρθεί. Και σας υπέσχομαι ε, επίσημα ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Σας παρακαλώ κυρία Άστον μην απαντήσετε σε μένα αλλά σε αυτούς σας κοιτούν. Όπως θα μας κοιτούν και πάντοτε με απορία διότι πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή την ανθρωπιστική τους αποστολή. Ε, όλοι καταδικάζουν την ε, ε, επιδρομή και ζητούν την άρση της, του αποκλεισμού αλλά δεν πρέπει να το ξεχάσουμε διότι θα υπάρξουν οι εκατοντάδες των συμμετεχόντων στο σχολείο του Μαρμαρά που θα έρθουν να μας το υπενθυμίσουν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 μια σκέψη στα θύματα του στόλου των ειρηνιστών, αλλά και μια σκέψη για το Ισραήλ. Ε, κυρίως σήμερα που η ολόκληρη διεθνής ε, κοινότητα ή σχεδόν ε, το κοιτά επικριτικά. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα λέω ότι στο κράτος του Ισραήλ θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα αιτιολόγησή του και ότι ο διάλογος δεν θα πρέπει να διακοπεί. Γιατί αν σβήσει αυτή η αγωνία για την ασφάλεια αλλά και για την δημόσια κοινή γνώμη αυτής της χώρας που αισθάνεται ανασφαλής, το καταλαβαίνουμε. Αλλά εμεί θέλουμε και την ασφάλεια και του Ισραήλ και την ευημερία του και την ηθική του ευημερία. Και γι' αυτό ακριβώς η επιθυμία να ακούσουμε τα αίτια του Ισραήλ κινείται από την ανώτατη επιθυμία της ειρήνης και από την, το καθήκον να πούμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι εδώ και χρόνια δεν καταλαβαίνουμε πια την πολιτική του. Όσα συνέβησαν δεν είναι ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που συνδέει ε την ε, την ε, επίθεση κατά του Στολίσκου με την απέλαση των ε, Αράβων, την κατασκευή των, ε, του τείχους, ακόμα και η άσχημη αυτή, η στάση του Ισραήλ απέναντι στους Άραβες της περιοχής. Είναι μια ταπεινωτική πολιτική που καθιστά πιο έντονο στους εξεμισμούς από όλες τις πλευρές, ακόμα και από πλευράς του Ισραήλ, απομακρύνοντας πάντοτε για πάντα ίσως την πιθανότητα, την προοπτική για μια ε, για τη δημιουργία δύο κρατών ε, που θα ζουν ειρηνικά πλάι-πλάι. Είναι ένα μια κόκκινη γραμμή πάνω στην, οποία, πάνω στην οποία κινείται ολόκληρη η πολιτική. Αλλά η τραγωδία αυτού του στολίσκου ε, θίγει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Με αυτό το με αυτές τις επικίνδυνες πολιτικές αποκλήσεις. Το ψήφισμα που έχουμε σήμερα καλεί στην πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική, ειδικά σήμερα που έχουμε κάποιες θεσμικές δυνατότητες. Δεν έχουμε πλέον δικαιολογίες ε, για να φωνάξουμε δυνατά, να ακουστεί η φωνή μας. Ε, δεν θα πρέπει να χαρακτηριστούμε απάνθρωποι. Τουλάχιστον οι πολιτικές μας θα πρέπει να μην είναι απάνθρωπες. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε πρόσωπε, νομίζω ότι εδώ στη Μικύκλιο συμφωνούμε όλοι, καταδικάζουμε όλοι την επίθεση στο Στολίσκο που προσπαθούσε ουσιαστικά να άρει τον αποκλεισμό της Γάζας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε με το ότι η Ισραηλινή πολιτική ως έχει αυτή τη στιγμή όπως υλοποιείται, επαναλαμβάνοντας αυτά που κάνει εδώ και χρόνια, ουσιαστικά οδηγεί το ίδιο το Ισραήλ ε, σε μία τρύπα από την οποία πολύ δύσκολα θα βγει. Όλοι συμφωνούμε. Το θέμα όμως είναι τώρα. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική αυτή. Το είπατε και εσείς οι ίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την συμφιλίωση, αν θέλετε, για την επίτευξη μια συμφωνίας μεταξύ των Παλαιστινιακών φρατριών εσεί, α πούμε δυνάμεων. Εγώ προτιμώ αυτόν τον όρο. Από την άλλη πλευρά, είτε μα αρέσει είτε όχι, υπάρχει αυτή η ε, κατάσταση Εμένα δεν μ' αρέσει που έχουμε τη Χαμάς και όχι την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά αυτό υπάρχει. Ω πολιτικοί πρέπει να δεχθούμε την πραγματικότητα και α μην μα κάνει να ονειρευόμαστε. Επομένω. πρέπει να έρθει ο υποκλεισμό και ο διανοητικό αποκλεισμό όμω που ε, έχουμε εμεί εδώ, ίσω έχουν και οι Ισραηλοί, ίσω έχουν και οι Παλαιστίνοι. Προτείνω λοιπόν το εξή. Είπατε, είπατε ότι πρέπει να αρθεί ο αποκλεισμό. Όχι μόνο στη Ράφα, όλα τα σημεία διέλευσης πρέπει να ανοίξουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και ζητεί να δει έλεγχοι. Τι έλεγχοι μπορούν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσε και ο τουρκικός στρατός να βοηθήσει. Ξέρετε ότι οι Γερμανοί και οι Τούρκοι στρατιώτες, αυτό είναι ηρωνία, ε, θα μπορούσαν να ελέγχουν ε, την είσοδο στη Γάζα ώστε να μπορούν να μπαίνουν τα τρόφιμα, να μπορούν να μπαίνουν ε, τα υλικά, τα δομικά για την ανοικοδόμηση τη χώρα κτλ. Ας χρησιμεύσουμε κι εμείς λοιπόν, α μην ζητούμε απλά να ανοίξουν τα σημεία διέλευση και να έρθει ο αποκλεισμό α το κάνουμε κι εμεί. Τώρα θα μπορούσα, αν μου επιτρέπετε, ε, να πω κάποια πράγματα στα γερμανικά, διότι πολλοί στη Γερμανία και στην Ευρώπη έχουν ένοχη τη συνείδησή τους ε, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Αλλά όταν έχει κανείς, θέλει να έχει ήσυχη τη συνάδεσή του και να βοηθήσει το Ισραήλ, πρέπει να πούμε στο Ισραήλ ότι αυτό που συμβαίνει τώρα ξεπερνά τα όρια του αποδεκτού. Οι φίλοι του Ισραήλ είναι οι κατακριτές του. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατακρίνουν τώρα το Ισραήλ δεν είναι φίλοι του. Και γι' αυτό άνθρωποι όπως ο Ντάβιτ Ρόσμαν ο οποίος πολύ σωστά είπε στο Ισραήλ ότι αυτό το οποίο έκανε το Ισραήλ ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον αντιλέγει ουσιαστικά το λόγο για τον οποίο ιδρύθηκε το Ισραήλ. Η πολιτική αυτή είναι μία ε, πολιτική η οποία δεν υλοποιεί το σιωνιστικό όνειρο αλλά το καταστρέφει. Άρα εμείς σαν Ευρωπαίοι δεν πρέπει να φοβόμαστε την κριτική έναντι των ε, Ισραηλινών και έναντι των ε, Παλαιστινίων. Ναι, χρειαζόμαστε μία νέα σταθερότητα στην περιοχή και αυτή θα επιτευχθεί μόνο εάν εμείς σαν Ευρωπαίοι είμαστε έτοιμοι να σταθούμε σταθούμε στη μέση σαν μία δύναμη η οποία θα είναι διαμεσολαβητής αλλά και ρυθμιστής. Αν δεν το πράξουμε αυτό δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε τάξη ούτε ρύθμιση. Γι' αυτό και σας παρακαλώ όχι μόνο να κάνετε κλήσεις να διατυπώσετε προτάσεις πώς εμείς οι Ευρωπαίοι με την Τουρκία που είναι σημαντική σε αυτή την περιοχή μπορεί να συμβάλλει για να αναλυφθούν συγκεκριμένα βήματα και να λήξει αυτός ο αποκλεισμός και σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Βαντάλεν. Για ένα λεπτό. Er Πρόεδρε, στις 31 Μαΐου, 9 νεκροί έπεσαν μετά από την παρέμβαση του Ισραήλ στα σκάφη στην ε, θάλασσα του Μαρμαρά. Τα σκάφη αυτά ε, Οι Ισραηλινοί λένε πως ε, δεν είχαν καλή υποδοχή στα σκάφη γιατί αναγκάστηκαν να αντιδράσουν. Ε, ε, δεν ξέρω τι μπορεί να περίμεναν, τσάι και γλυκά. Και γι' αυτό και το μέγα ερώτημα είναι γιατί το Ισραήλ δεν, δεν σταμάτησε τα σκάφη με άλλα μέσα. Υπήρχαν άλλες επιλογές για τον Ισραηλινό στρατό που δεν θα είχαν ε, τόσα θύματα και θα είχαν οδηγήσει σε πολύ λιγότερη βία. Είναι λοιπόν απόλυτα θεμητό να γίνει έρευνα και το Ισραήλ αντέδρασε με θετικό τρόπο. Θα γίνει έρευνα με την εμπλοκή δύο διεθνών προσωπικότητων. Καλύτερα είναι να γίνει ο κατάλογος των πραγμάτων που δεν μπορούν να μπουν στην Γάζα. μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το πρωινό της 31 Μαΐου ο Ισραηλινός στρατός επιτέθηκε από αέρα και θάλασσα στο στολίσκο της Ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστικό υλικό στους κατοίκους της Γάζας σκοτώνοντας άνανδρα εννιά ακτιβιστές και πληγώνοντας δεκάδες άλλους μερικοί εκ των οποίων μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή από τον εξώστη. δεν είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προβαίνουν σε εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας. για 23 συνεχόμενες μέρες και νύχτες σφυροκοπούσαν ανελέητα τη γάζα στην οποία βρίσκονταν αποκλεισμένοι πυκνοκατοικούντες 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι Προκαλώντα το θάνατο σε 1.400 καταστρέφοντα την ηλική υποδομή και αφήνοντα πίσω του και αποκαΐδια. μήπω αναγκάστηκαν να λογοδοτήσουν για, αυτό το έγκλημά του σε κανένα. Καθημερινά οι κατοχικέ δυνάμεις υποσκάπτουν τι διεθνεί προσπάθειε για εξέβρεση λύση σε ένα πρόβλημα που οι ίδιες συντηρούν εδώ και έξι δεκαετίε. Συνεχίζουν να προεκτείνουν το διαιρετικό τείχος, να οικοδομούν νέου οικισμού επίκων, να διώχνουν από τα σπίτια τους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ φιλήσυχους Παλαιστίνιους. Μήπως αναγκάστηκε το Ισραήλ να λογοδοτήσει για αυτή του την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, αύριο θα κληθούμε να ψηφίσουμε ένα κοινό ψήφισμα καταδίκης της επίθεσης των Ισραηλινών στρατευμάτων ενάντια στο στόλο της ελευθερίας. Ας μην εφησυχάσουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο επιτελούμε το καθήκον οφείλουμε ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να εργαστούμε για να καταστούν οι ένοχοι υπόλογοι ενώπιον δικαστηρίου αλλά και για να αρθεί επιτέλους αυτός ο απάνθρωπος αποκλεισμός της γάζας και για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή. το οφείλουμε στους νεκρούς ακτιβιστές στα θύματα και των δύο πλευρών της πολύχρονης διένεξης στους λαούς του ισραήλ και της παλαιστίνης. Εξ ονόματος Ευρώπης και Δημοκρατία, ο κύριο Μπέλντερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ε, την τουρκική κυβέρνηση ε, και το Ίδρυμα, ε, το τουρκικό για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε να ξεχάσουμε την αποτρόπα επίθεση των Ισραηλινών στο στόλο της ελευθερίας. Γιατί κανείς δεν μίλησε, γιατί και εσείς κυρία Ήπατη εκπρόσωπε τηρήσατε σιγή. Κυρία Άστον, Γνωρίζετε κι εσείς ε, ποιος ε, εκρυβόταν πίσω από το στολίσκο αυτό της ε, ελευθερίας. Είναι μια ανθρωπιστική βοήθεια κάπως ιδιόμορφη ουσιαστικά που έχει κάποιες άλλες δράσεις και ξέρουμε τι είχε πει και ένα ηγετικό της τέλεχος πέρυσι μέχρι είχε μιλήσει και για Τούρκο μάρτυρα. οι τουρκικές αρχές μετά από αυτό το δράμα βέβαια που συνέβη, αυτή την τραγωδία, ζήτησαν ε, ε, το λογαριασμό από το Ισραήλ. Εμείς τι κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για το πλοίο ε, Μαρμαρά. Κυρία, είπατε, είπατε εκπρόσωπε, πρέπει επίσης ο στρατιώτης ο Ισραηλινός να απελευθερωθεί. Πρέπει κάτι να γίνει και γι' αυτό. Ευχαριστώ. μία η κυρία Ντότζ για ένα λεπτό. Thank you, uh, Mr. President, uh, Baroness Ashton. Um, Πρόεδρε, κυρία Άστον, ε, χαιρετίζω την δήλωσή σας και θυμάμαι την πρώτη σας δήλωση σχετικά με το Ισραήλ και την Γάζα και αναγνωρίζω ότι τώρα είναι πιο μετριασμένη και πιο πλήρης η δήλωσή σας όπως είπε ο συνάδελφός μας. Για όσους από εμά έχουν ζήσει ε, τρομοκρατικές απειλές ε, καταλαβαίνω απολύτως τους πολίτες οι οποίοι του Ισραήλ οι οποίοι υποφέρουν ε, από ανεξέλεγκτες, ε, ε, ανεξέλεγκτους πυράβλους και η κατάσταση στη Γάζα κάπως μείωσε τους κινδύνους του Ισραήλ και άρα ο καθένας δικαιούται να προστατεύσει το λαό του από τέτοιες επιθέσεις. Για το λαό της Γάζας δημιουργήθηκαν δυσκολίες και αντιλαμβάνομαι ότι ότι πολλοί θα σηκωθούν υπέρ του στολίσκου της ειρήνης αλλά υπήρχαν και άτομα των οποίων οι προθέσεις δεν ήταν τόσο ευγενείς και υπήρχε μία προσπάθεια δημιουργίας αντιπαράθεσης και τυχώς είχαμε απώλειες ζωής θα, με αυτόν τον τρόπο προχωρήσαμε τη συζήτηση για το Ισραήλ εδώ, αλλά αυτό δεν βοηθά την Ιρίζη Νομίζω ότι ξεπεράσατε την ώρα σας. Μπορεί όμως να μένουν στην ε, φυλακή ε, ένας όμηρος πέραν των 1400 ημερών για αυτό το λόγο. Για 1,5 λεπτό. Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους εγγραμμένους ομιλητές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε ανθρωπιστικό στολίσκο ή στρατηγική πρόκληση. Ε, ακούμε αντιφατικά ε, σχόλια. Θα πρέπει όμω να εκφράσουμε τη λύπη μα για τη χρήση βία από πλευρά Ισραηλινών αλλά και τη λύπη μα για την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Και για όλα αυτά υπάρχουν αίτια τα οποία οδήγησαν σε κάποιε συνέπειε. Πέραν του πλέον οδυνηρού που είναι όπω είπα η απώλεια ανθρώπινων ζώων είναι επίσης ε, και η εξάρθρωση τη ειρηνευτική διαδικασία, η απομόνωση του Ισραήλ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι ΗΠΑ, οι κακέ σχέσει με του ε, με τις ε, μετροπαθείς αραβικές ε, χώρες. Έχουμε επίσης το, το πυρηνικό, την πυρηνική απειλή του Ιράν να πλανάται στην ατμόσφαιρα και όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Η κυρία Άστον είπε κάτι που με βρίσκει απόλυτο σύμφωνο. Το να ε, δώσουμε στον ε, Παλαιστινιακό λαό πίσω την αξιοπιστία του αυξάνοντας ε, τις, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής του σίγουρα είναι υπέρ και των μετριοπαθών και της Ένωσης και της, του Παλαιστινιακού λαού και σίγουρα η άρση του αποκλεισμού γι' αυτό είναι μόνο ένα βήμα προς αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε την αναγνώριση ενό βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτου. Θέλουμε να υπάρχει ασφάλεια στα σύνορα του Ισραήλ. Θέλουμε να λυθεί το ζήτημα τη Ανατολική Ιερουσαλήμ, το ζήτημα των επικισμών που πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα και ολοκληρώνω. Για να λύσουμε το Παλαιστινιακό, δύο λύσει. Το πρώτο είναι η πολιτική βούληση και το δεύτερο είναι η ε, παρακολούθηση εκ μέρου τη διεθνού κοινότητα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτική βούληση απαραίτητη τουλάχιστον στο βαθμό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος για ένα λεπτό. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμά μας είναι ξεκάθαρο στην καταδίκη των παράνομων πράξεων του Ισραήλ που σκότωσαν 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν 28. Ε, Θέλουμε έρευνα διεθνή, διαφανή και ανεξάρτητη. Η έρευνα από πλευρά του Ισραήλ δεν είναι κανένα από αυτά τα πράγματα και δεν είναι αποδεκτή. Εμείς θέλουμε το τέλος του αποκλεισμού της Γάζα. Πιο σημαντικό παράγραφος είναι η 10 του ψηφίσματος που ζητά την, ε, τον μετασχηματισμό της πολιτικής της Ένωση προ την Μέση Ανατολή και αυτό θα πρέπει να περικλεί το διπλωματικό εργαλείο των κυρώσεων αφού το Ισραήλ δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφέ ενό δημοκρατικού κράτου ε, στην ε, αντιμετώπιση των φίλων και των εχθρών του. Θα πρέπει λοιπόν ε, λήψη αντίδραση από το Ισραήλ να σεβαστεί τη, διεθνή, τη, το, διεθνή νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξουν κυρώσει. Ε, δεν είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε συμφωνία δύο κρατών χωρίς τη συμμετοχή και των δύο στη διαδικασία. Ο πιο δημοκρατικός τρόπος να προχωρήσουμε είναι να γίνουν ε, εκλογέ στην Παλαιστίνη και για τον πρόεδρο τη Παλαιστινική Αρχή με τη συμμετοχή όλων αλλά και από το κουαρτέτο ώστε να αποδεχτεί την απόφαση του λαού. Πρέπει να ενεργήσουμε πια. Η κυρία για ένα λεπτό. Euh, το διαπιστώσαμε επί τόπου ότι οι κάτοικοι εξαρτώνται κατά 80% από τη διεθνή βοήθεια. Δεν ζουν, επιβιώνουν χωρίς μέλλον και χωρίς καμία ελπίδα. Ο αποκλεισμό της ε, Γάζας απλώς δίνει ε, αυτό που θέλει κανείς να αποφύγει και ε, δίνει τη δυνατότητα εις τους ηθήνοντες της Γάζας να δικαιολογήσουν τα πάντα. Πρέπει λοιπόν λοιπόν η Ευρώπη να δράσει και να εγγυηθεί την ε, ασφάλεια του Ισραήλ, να εξασφαλίσει την κατάργηση του αποκλεισμού ενδεχομένως με ευρωπαϊκό έλεγχο. Πρέπει να λειτουργήσει με μία μόνο φωνή και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα πολιτικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά για να εξυπηρετήσει ένα μόνο στόχο, τη μακροπρόθεσμη συνύπαρξη δύο κρατών. Ευχαριστώ. Madame la Haute Représentante et chers collègues. Κυρία είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την επίσκεψή μας ε, στην ε, Γάζα 26 με 27 Μαΐου ήταν ομόφωνη η ε, έκκλησή μας ε, για διαρκή μόνιμη άρση του αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Γάζα το Ισραήλ. Λαμβάνοντα υπόψη αυτό το δράμα, αυτή την ε, τραγωδία, την ανθρώπινη και πολιτική, αυτό το κοινό ψήφισμα το οποίο έχουμε υποβάλει, ελπίζω να εγκριθεί ομόφωνα γιατί θέλουμε να εκπέμψουμε ένα και νέο μήνυμα. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό, διότι ουσιαστικά ε, αυτό που έλειπε μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η ενότητα και αυτό χρειαζόμαστε για να βαρύνει η άποψή μα, ε, για να βαρύνει ο ρόλο μας ε, ως ένα σημαντικός ειρηνευτικό παράγοντας. Ας μην προσθέσουμε στο δράμα, στην τραγωδία του Στολίσκου, την άγνοια και την, την μα και την παραγνώριση των προβλημάτων δεν έχουμε μόνο δικαίωμα, έχουμε το καθήκον να δράσουμε, να ε, διαλεγούμε και βέβαια και να τιμωρήσουμε, να ε, κολλάσουμε όταν βλέπουμε να παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα ότι από την άλλη πλευρά. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι, έχουμε τεράστια ευθύνη σήμερα. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε πλέον στην ε, ανοικοδόμηση ενό συμπλέγματο κτηρίων. Την ειρήνη πρέπει να επαναφέρουμε και αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Και αυτό απαιτείται βέβαια και σταθερότητα, επιμονή και σθένος πρέπει να ε, συμπήξουμε συμμαχίες, ε, όχι μόνο με την Τουρκία. Θα πρέπει ε, να επιβάλλουμε κάποιους όρους στο Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές σχέσεις μέχρι ότου αρθεί πλήρως ο αποκλεισμός. Ο κύριος Καρίμ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε, σας συγχαίρω, Βαρονιά, για τον τρόπο με τον οποίο προσχεδίσατε το το, την κατάσταση αυτή ε, και η επίσκεψή σας διευκρινίζει με πόσο σοβαρότητα έχετε προσεγγίσει το θέμα αυτό. Είναι βέβαια ένα θέμα ανθρωπιστικό μαζί με πολλά άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν. Αλλά αν κοιτάξουμε την ιστορία θα δούμε γιατί βρισκόμαστε όπου βρισκόμαστε τώρα. Και θυμάμαι ότι έχουν γίνει συζητήσεις εδώ το 2006 και το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο όπου πάρα πολλοί ευρωβουλευτές είχαν κάνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ να μην αποκλείσουν έτσι το λαό της Γάζα και κάναμε ακριβώς αυτό. Η αντίδρασή μας ήταν λαθασμένη. Τους αποκλείσαμε και τώρα μπορούμε μόνο να λύσουμε το θέμα εάν αντιμετωπίσουμε τον αποκλεισμό απευθείας και να λάβουμε μέτρα εκ των οποίων το πρώτο θα είναι να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ θα λειτουργήσει με τρόπο που θα επιτρέπει επιτρεπόμενα εμπορεύματα να περνούν και όχι μόνο με ένα ε, κατάλογο όπως γίνεται τώρα και παρακαλώ να εστιάσετε την προσοχή σε αυτό το θέμα αμέσως. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Εδώ και υπερβολικά πολύ καιρό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν τα ίδια ευχολόγια με καλές προθέσεις που διακηρύσσονται χωρίς να αναλαμβάνονται ενέργειες για την ειρήνη στην περιοχή και ε, για την ύπαρξη ε, ενός παλαισιακού καράτους στα όρια του 1967. Έγινε είναι πειρατεία από πλευράς διεθνούς δικαίου σε μια ανθρωπιστική νιοπομπή. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν την ε, έρευνα να την κάνει ο ίδιος ο δράστης για να μας ικανοποιήσει ούτε καν με ε, ένα ασαφές πρόγραμμα μειώσεως αυτού του αποκλεισμού που θα ικανοποιηθούμε. Πρέπει να απαιτήσουμε την πλήρη άρση του αποκλεισμού. Έχετε μέσα, ας δημιουργήσουμε αποστολές ε, ευρωπαϊκής εποπτείας σε συνεργασία με άλλα κράτη ε, στα σημεία διελεύσεως από και θαλάσσης και να μην υπάρχει, ε, ε, ε, να υπάρξουν ποινές κατά του Ισραήλ όσο δεν γίνονται βήματα, να σταματήσει η συνεργασία στα θέματα στρατιωτικής τεχνολογίας και να πάψουν οι πωλήσει όπλων στο Ισραήλ. Και θέτω το ερώτημα, ποιος θα εξετάσει τους ξυλοδαρμούς των Ευρωπαίων τις ε, φυλακέ του Ισραήλ. Ε, θα ζητούσα ε, κυρία κυρία Επίτροπε να προχωρήσετε με τις σωστές ενέργειες και θα σας στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Από μια πρώτη επαλήθευση των γεγονότων ε, είναι προφανές ότι η αποστολή του Στολίσκου στη Γάζα είχε στόχους περισσότερο πολιτικούς παρά ανθρωπιστικούς. Ε, η αποστολή προετοιμάστηκε από την ε, IHH, μια τουρκική οργάνωση που συνδέεται με τον Ισλαμικό Εκστρεμισμό. Επιπλέον την προηγουμένη της αναχώρησης του Στολίσκου, ο αρχηγός της Χαμάς Ανιέ δήλωσε συγκεκριμένα αν τα σκάφη φτάσουν στη Γάζα θα είναι νίκη για την Χαμάς. Αν αναχαιτιστούν θα είναι και πάλι νίκη. Το μικρό ενδιαφέρον όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς στόχους αυτής της αποστολής επιβεβαιώνεται από την άρνηση της Χαμάς να, να δεχτεί στην Γάζα την ανθρωπιστική βοήθεια που φτάνει μέσω του λιμανιού Ασχόντ με το ε, σκάφος Ρέτσελ Κόρι. Αν νικήσει η Αμάς δεν χάνει μόνο το Ισραήλ αλλά και η Παλαιστινιακή Αρχή και η δυνατότητα να ξαναρχίζει η, διαδικασία, η ειρηνευτική διαδικασία η, θαλάσσια και η χερσαία, ο θαλάσσιος και χερσαίος αποκλεισμός στην Γάζα που έχει επιβάλει το Ισραήλ και η Αίγυπτος από το 2007 για να ελεγχθεί το εμπόριο όπλων έγινε δεκτό πριν από λίγες μέρες από τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντα Μπάς στην επαφή του με τον πρόεδρο Ομπάμα και αυτό το επιβεβαιώνουν όλες οι εφημερίδες. Δεν θα πρέπει η Γάζα να γίνει μια θέση, ένα θέατρο πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ και ένα στοιχείο αποσταθεροποίηση ε, στην ολόκληρη την περιοχή. Θα πρέπει ωστόσο να μπορέσει να υπάρξει δίωδο για την ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να ανακουφιστεί ο πληθυσμό τη Γάζα. Ζητώ από την είπα το εκπρόσωπο να επεκτείνει την έρευνα στα γεγονότα και στην πιθανή εμπλοκή χωρών όπω η Τουρκία και το Ιράν στην διοργάνωση τη αποστολή αυτή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάφορα εργαλεία και διάφοροι άνθρωποι που αυτοανακηρύσσονται οι υπερασπιστές της ειρήνης ε, μπήκαν στην πορεία για τη Γάζα. Ακούσαμε ένα σωρό πράγματα όσον αφορά την ε, ε, υποδοχή των ανθρώπων του Ισραήλ που έφτασαν στα σκάφη, αυτή έγινε με ρόπαλα και με μεταλλικές ράβδους. Οι επιβάτες των σκαφών δήλωσαν ότι υπήρχαν επαφές με τον Πρωθυπουργό Ερντογάν της Τουρκίας και ότι η κυβέρνηση της χώρας αυτής ήταν εμπλεγμένη στην προετοιμασία του στόλου αυτού. Είναι προφανές πως ε, ε, όλα αυτά είναι συνδεμένα με την ΑΜΑΣ, η οποία θεωρείται ε, τρομοκρατική οργάνωση. Θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον μια ανεξάρτητη έρευνα για το ρόλο της Τουρκίας σε όλα αυτά. Ποια ήταν η επιρροή του Ερντογάν σε όλη αυτή την υπόθεση. vielen Dank, Herr Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, στηρίζω την απέτηση για μία διεθνή έρευνα και τη συμμετοχή δύο διεθνών εμπειρογνωμόνων εις ε, την ε, στην Ισραηλινή έρευνα διότι αυτή δεν επαρκεί ε, για να δούμε αν ήταν παράνομες οι δράσεις αυτές και μέχρι τότε νομίζω ότι θα έπρεπε να περιορίσουμε τις αξιολογήσεις μας. Μία τέτοια, ένα τέτοιο στολίσκος μπόρεσε ε, να, ε, να ξεκινήσει και δεν περιείχε μόνο αντιδραστικά στοιχεία για ανθρωπιστικό στόχο και ε, το, ούτε το Ισραήλ επέτυχε το στόχο του ούτε ε, το Χαμάς διότι ε, δεν, δεν εστράφησαν κατά του Χαμάς οι κάτοικοι της Γάζα αλλά κατά του Ισραήλ και ο Όμηρος δεν απελευθερώθηκε. Ελπίζω λοιπόν ότι σήμερα θα μπορέσει μπορέσει να ισχύσει η απόφαση ότι θα χαλαρώσει ο αποκλεισμός και θα υπάρξει μια σχετική απελευθέρωση σε ορισμένα εμπορεύματα τα οποία δεν είναι όπλα ή υλικά με τα οποία μπορεί να κατασκευάσει κανείς οπλισμούς. Θα έπρεπε επίσης το Ισραήλ να σκεφτεί εάν η πρόταση των Γάλλων και των Βερτανών που διατυπώθηκε χθε μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή ε, να ελέγχονται τα πλοία τα οποία ε, πηγαίνουν προς τη Γάζα. Grazie, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα όσα συνέβησαν. Και θα ήθελα να πω ότι βρεθήκαμε ενώπιον μιας πράξης ε, βίαιης Ε, βίες επιθετικότητα από πλευράς του Ισραήλ. Ίσως ε, θα πρέπει να γίνει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες ώστε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία και όχι τέτοιου είδους ε, ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μια σημαντική ε, απάντηση από πλευράς μας για το δύσκολο θέμα της Γάζας. Ωστόσο αυτή η δραματική ενέργεια απαιτεί από την Ευρώπη ένα ποιοτικό άλμα στην αντιμετώπιση της, του Μεσανατολικού. Κυρία Άστον, πιστεύω πως εσείς γνωρίζετε πως σήμερα χρειάζεται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο νέο τύπο η Ευρώπη, μια πιο έντονη δράση θα έχει ως στόχο να ξαναβάλει στο σωστό δρόμο τις ε, διαπραγματεύσεις, να σταματήσει αυτή η πολιτική των, ε, ε, ε, του επικισμού και να περιοριστεί ή να καταργηθεί και τελείως ο αποκλεισμός της Γάζας. Να μην αναφέρεται καμία... Θα πρέπει μάλλον κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστεί η σύγκρουση και να ετηθούν οι εξτρεμιστικές δράσεις που είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν και τα δύο κράτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα ε, θύματα της 31 Μαΐου αξίζουν ε, την εκτίμησή μας και πρέπει να τους θυμόμαστε. Ε, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε λανθασμένη πολιτική. Οι ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν ήταν μόνο ατυχής αλλά δεν ήταν άξιες ενός συγχρόνου κράτους κράτος δικαίου. Υπάρχει πέραν του φυσικού αποκλεισμού και ένας πολιτικός αποκλεισμός στην Ιερουσαλέμ και ε, ε, υπάρχει τελείως λάθος εκτίμηση των κινήσεων αυτό. Έπρεπε λοιπόν η Επιτροπή να είναι διεθνής, δεν θέλει να υπάρξει μία δεύτερη Επιτροπή Goldstone 2, θα πρέπει να ανοίξουν τα ε, σύνορα με πιο σταθερή εντολή αν ε, θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε και πάλι σαν Ευρωπαίοι. Είναι όμως βασικό να ε, επηρεάσουμε το Χαμάς, να σταματήσουν οι εκτοξεύσεις πυράβλων και να απελευθερωθεί ο Ισραηλινός Όμηρος. Κυρία Φλότχα, για τα νέα θύματα από το στολίσκο της ελευθερίας ε, που δέχθηκαν ε, σχεδόν ε, εξ επαφής και κάποιες φορές πισόπλατα πάρα πολλές σφαίρες μπορεί να είναι ίσως όχι τόσο σημαντικό ποια εθνικότητας είναι όμως τουρκικής εθνικότητας παρόλα αυτά και ίσως σήμερα κάποιοι θέλουν μετά από όλες αυτές τις δράσεις, αντιδράσεις και πιέσεις ε, που ασκεί στην Ισραηλινή κυβέρνηση η κυβέρνηση Ερντογάν θα θέλαν να βάλουν ε, το στίγμα του ότι πρόκειται για μια Ισραηλοτουρκική υπόθεση. Θα μπορούσε δηλαδή να θεωρηθεί ότι πλέον ε, αλλάζει πλεύση η, Τουρκία και στρέφει την πλάτη της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να πούμε ε, κυρία Άστον ξεκάθαρο ότι ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή πολύ καλά δέχεται τα συγχαρητήρια των ε, μουσουλμάνων ηγετών διότι ουσιαστικά διοπραγματεύεται και αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το ριζοσπαστισμό και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τον υποστηρίξουμε και να τον ενθαρρύνουμε και σας ζητώ να το κάνετε αυτό κυρία Άστον ξεκάθαρα κιόλας. Ο κύριος για 1,5 λεπτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταδικάζει με αποτροπιασμό και αγανάκτηση την εμψυχρό δολοφονική επίθεση του Ισραηλινού στρατού κατά της νιοπομπής αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες που συγκλώνησε τους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η νέα αυτή θηριωδία του Ισραηλινού κράτους αποτελεί κρίκο στη μακριά αλυσίδα των εγκλημάτων του Ισραήλ που έχει πάρει διαστάσεις γενοκτονίας ενάντια στον παλαιστινιακό λαό. η προκλητική στρατιωτική δράση του ισραηλινού κράτους στηρίζεται και πρημοδοτείται σταθερά από τις Ηνωμένε Πολιτείε της αμερικής το νατο και την ευρωπαϊκή ένωση καθώς και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. σοβαρές ευθύνε έχουν η ευρωπαϊκή ένωση και οι κυβερνήσει των κρατών μελών τη, που όχι μόνο ανέχονται την ισραηλινή επιθετικότητα που όχι μόνο αναβάθμισαν τις σχέσεις τους με το ισραήλ υπέγραψαν τη δημιουργία ενιαίου εναέριου χώρου με την ισραηλινή κυβέρνηση και συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας αλλά και διοργανώνουν μεγάλης έκτασης κοινά στρατιωτικά γυμνάσια τροφοδοτώντας την εγκληματική επιθετικότητα του ισραήλ σε βάρος του παλαιστινιακού λαού και γενικότερα σε βάρος των λαών της ευρύτερης περιοχής η συγκρότηση της ερευνητικής επιτροπής για την αιματερή επίθεση του ισραηλινού στρατού στην ιοπομπή βοήθεια προς τους κατοίκους της γάζας που συνέστησε στα μέτρα της η ισραηλινή κυβέρνηση προκλητικά εξήγηλε ότι στόχος της είναι να διαφυλάξει την ελευθερία δράσης των ισραηλινών στρατιωτών και να αποδειχθεί ο αμυντικός χαρακτήρας των ενεργειών τους δηλαδή να δικαιολογήσει και να συνεχίσει τις δολοφονικές επιθέσεις της ενάντια στον παλαιστινιακό λαό και στους λαούς της ευρύτερη περιοχής γι' αυτό και οι εκκλήση της ευρωπαϊκής ένωσης για σύσταση δήθεν ανεξάρτητη διευθυντική επιτροπής αποτελούν κοροϊδία και υποκρισία. ο Παλαιστινιακό λαό δεν έχει ανάγκη από διερευνητικές επιτροπέ που θα συσκοτίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα σε βάρο των παλαιστινίων. τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η αντιπεριαλιστική πάλι των λαών να δημιουργηθεί ενιαίο ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να διακόπτω. Ξέρω ότι είναι ενοχλητικό το σφυρί. Ελπίζω ότι όσοι το ακούτε θα σταματάτε σχεδόν αμέσω για να μπορέσουμε να, να κρατήσουμε το χρόνο. Ε, η κυρία Τζαβέλα για 1,5 λεπτό. Πρώτα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά λύπη μου για τους θανάτους που είχαμε σε μέλη της νιοπομπής. Παράλληλα όμως κάνω έκκληση κυρία Άστον προς όλους σας να μην παρασυρθούμε από αυτό το δυστύχημα για να εξάγουμε μια αντικειμενική θεώρηση των πραγμάτων. λυπάμαι αλλά στη μέση ανατολή θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς τα αγνά κίνητρα των ακτιβιστών. θα έλεγα ότι πολλές φορές έχουμε δει επιδίωξη δημιουργίας μαρτύρων παρά ακτιβιστική δράση προσωπικά επίσης εκφράζω την έκπληξή μου για την ύπαρξη μιας πολύ καλά οργανωμένης ακτιβιστικής τουρκικής οργάνωσης με όλο το σεβασμό στα μκο της τουρκίας δεν νομίζω ότι φημίζεται η τουρκία για την ελευθερία ε, του ακτιβισμού αυτών που θέλουν να είναι ακτιβιστές. για όλα αυτά κυρία άστον και για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα των πραγμάτων. θα παρακαλούσα να συστήσετε μια επιτροπή διερεύνησης των δράσεων και του ιστορικού της ανθρωπιστικής οργάνωσης ihh. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Μέλτσερ, για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, να τα ισχύει αυτό το οποίο είπε ο κύριος Προβέρα και Μπέλτερ. Δηλαδή ότι υπήρχαν ε, και προκλητικές ισλαμιστικές δυνάμεις πίσω από τον στολίσκο της Γάζα και πρέπει να ξέρει κανείς πώς τοποθετούνται. Αλλά ε, η επίθεση από τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς είναι μία πράξη βίας και ε, νέα σκοτώθηκαν και ε, άλλοι ε, είχαν ε, τραυματιστεί. Πρέπει λοιπόν κανείς να μειώσει τις, τις δράσεις αυτές και οι πράξεις αυτές των κομμάντων είναι η βάρος των εταίρων του Ισραήλ όπως η Ευρώπη οι οποίοι είναι δύσκολο να υπεραμεινθούν ενθούν της ε, υπάρξεως του Ισραήλ αλλά υπάρχουν ε, διεθνή πρότυπα τα οποία ισχύουν και για τους Παλαιστινίους και γι' αυτό το λόγο ο αποκλεισμός ε, της Γάζας από τον οποίο υποφέρει ο λαός και οι πολίτες της Γάζας πρέπει να σταματήσει το ταχύτερο και γι' αυτό καλό τους υπευθύνους να αντιπροσωπεύσουν αυτή την την άποψη διότι υπάρχει μία μείωση των προσπαθειών για την ειρήνευση της Μέσης Ανατολής και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας θα πρέπει να συμβάλλει και το Ισραήλ. Ναι κύριε Πρόεδρες, ε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπη, καταρχήν θέλω να ε, εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των ε, ατόμων και να καταγγείλω την επιδείνωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης, υπερβολικός αριθμός ανέργων και υποσυτιζομένων. Η εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια και μόνο. Η αρχή αυτή της ε, ανθρωπιστικής ε, κινήσεως πρέπει να αναλάβει μέτρα για να σταματήσει η ισχύουσα κατάσταση. Είχα πάει στη Γάζα πριν δύο εβδομάδα, η κατάσταση των πολιτών είναι απαράδεκτη και οι πραγματικοί φίλοι του Ισραήλ είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή έχουν το θάρρος να καταδικάσουν το Ισραήλ για αυτό τον αποκλεισμό ο οποίος ε, δεν είναι άξιος του λαού του Ισραήλ. Πρέπει κυρία Άστον να σταματήσουμε αυτό τον αποκλεισμό και φτάνει λίγο θάρρος πολιτικό. Έχουμε τη δυνατότητα και τα μέσα να το επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ. κυρία Κρέτου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και είπατε εκπρόσωπε. Υπήρξαμε μάρτυρες ενός ε, πάρα πολύ τραγικού συμβάντος ε, με απώλεια ανθρώπινων ζώων. Φαίνεται ότι αυτή η βία δεν θα έχει ποτέ ένα τέρμα. Πάντως πρόκειται για κάτι καταστροφικό και για τον ειρηνευτικό διάλογο, τον συμφιλιωτικό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα από τη δική της πλευρά, ε, κυρία είπατε εκπρόσωπη, είναι ο σημαντικότερος χρηματοδότης στην περιοχή. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουμε και ο σημαντικότερος πολιτικός εταίρος Χρησιμοποιούμε μέτρα ε, πολύ σημαντικά, ε, αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε περισσότερα για να βοηθήσουμε τον Παλαιστινιακό λαό να βελτιώσουμε την, ε, τις συνθήκες διαβίωσης και θα πρέπει να έχουμε και έναν σημαντικότερο ρόλο και για την βελτίωση και την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα πρέπει να προαγάγουμε μια βιώσιμη λύση για, δύο, για τα δύο κράτη στην περιοχή. Ο κύριος Βάγκλ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Άστον, Μάλιστα. Όντως, ε, ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω με την παράκληση να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για να ε, θυμηθούμε τους νεκρούς. Αλλά δεν έχουμε ποτέ επαρκή χρόνο και ε, παρόλα αυτά θέλω να ε, ε, αναφέρω τους νεκρούς. Ευχαριστώ κυρία Άστον για την προσπάθειά σας και για τη διαπίστωση ότι έχει χάσει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν πιο ενεργό λόγο, ρόλο στη Μέση, Ανατολή, να εξασφαλίσει ότι θα γίνονται σε σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για όλους. Πολλοί μίλησαν για την λύση των δύο κρατών που θα συνυπάρχουν. Τι θα γίνει όμως ε, στην δυτική όχθη στην πραγματικότητα με αυτό. Δηλαδή ε, δεν θέλουμε να οξύνουμε το πρόβλημα της Γάζας διότι χρειαζόμαστε μια επιτυχή ε, αποστολή. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε, αυτή η τελευταία κρίση θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα σύμπτωμα των βαθιά δύσκολων σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης. Γιατί έχει σταθεί αδύνατο να βρεθεί λύση στη σύγκρουση ανάμεσά του. Η εύκολη απάντηση είναι ο ένα να τα ρίχνει στον άλλον, ότι είναι πιο υπεύθυνοι για όλα αυτά. Και οι δύο ομολογούν πω θέλουν ειρηνικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό που συμβαίνει όμω μα λέει άλλα είναι δεν είναι καθόλου προφανής ε, ότι μια λύση που θα είναι αποδεκτή για όλους θα είναι, είναι στο μυαλό των Παλαιστινίων ή των Ισραηλινών. Και οι δύο θεωρούν πως τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα από την σύγκρουση, γιατί οποιαδήποτε λύση θα κατέληγε στο να καταλήξουν σε πιο αδύναμη θέση από αυτή που κρατούν αυτή τη στιγμή. Ε, για, από την Ισραηλινή προοπτική επισήμω υπάρχει υποστήριξη για μια λύση των δύο κρατών, αλλά είναι δύσκολο να δει ένα Ισραηλινό κράτο θα συζούσε ειρηνικά με ένα Παλαιστινιακό κράτο, ε, Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε εξεπέραστα προβλήματα ασφάλειας. Από την άποψη της Παλαιστίνη, θα σήμαινε ότι αυτό θα έπρεπε εμά να, μην, να, να το μονοπόλιο της στην Γάζα και να το με την Φάτα. Ε, άρα λοιπόν μέχρι ότου του δοθούν κίνητρα ώστε να βρουν θέσεις καλύτερες από από ό,τι μέχρι τώρα η σύγκρουση τραγικά θα συνεχίζεται. Συνάδελφοι, κυρία Άστον, εγώ αντιπροσώπευα την, Επιτροπή Προπολογισμού στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Γάζα μία εβδομάδα πριν από τα τραγικά αυτά γεγονότα. Τουλάχιστον αυτά τα τραγικά γεγονότα μας ενώνουν σε κάποια συμπεράσματα και για μια νέα απο, ανανεωμένη προσπάθεια για την ειρήνη. Ε, ο αποκλεισμό σταματά την ανοικοδόμηση σπιτιών και σχολείων και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τη βοήθεια μέσω του ε, κοινοτικού προπολογισμού και άρα άμεση ευθύνη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω, έχει υπάρξει πάυση εργασιών λόγω έλλειψης υλικών στη διαδικασία νοικοδόμησης. Θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας. Η σημερινή κατάσταση όχι είναι μόνο πρόβλημα για τον αθώο πληθυσμό της Γάζα, περισσότεροι είναι παιδιά και νέοι, αλλά τροφοδοτεί τον εξτρεμισμό και την μαύρη οικονομία. Την παραοικονομία είναι απαραίτητο. Νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να διοργανώσει ειρηνικές μεταφορές στην Γάζα. I am a friend of... Είμαι φίλη του Ισραήλ, αλλά δεν θεωρώ ότι ε, ε, εάν κατακρίνουμε τις πράξεις τις τωρινές του Ισραήλ ε, χάνει κανείς την νομιμοποίηση του κράτους αυτού. Ε, πρέπει να σταματήσει ο αποκλεισμός ε, και δεν είμαι υπέρ της λύσης αυτής διότι δεν μπορούμε ε, πρώτα να καταδικάζουμε το Ισραήλ και μετά να ζητάμε μία διεθνή έρευνα και κάτι δεν είναι σαφές μεταξύ αυτών και η δράση του τουρκικού, της τουρκικής οργανώσεως Δεν φοβάμαι ότι η Τουρκία η οποία είναι θυμωμένη δεν μπορεί να ε, κυκλοφορεί φυλάδια ότι ο, ο ε, το Ισραήλ έχει χάσει την ομιμοποίησή του και ο σιωνισμός αποτρέπει τον, τον Ιουδαϊσμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει όντως ε, ε, να καταγγείλουμε και τα θύματα και τα στρα... τους ε, τραυματίες από τις στρατιωτικές πράξεις αλλά δεν πρόκειται απλώς για ανθρωπιστική προσπάθεια αλλά για ακτιβιστές διότι ο Στολίσκος αυτός πήγε εκεί τη στιγμή που ξαναξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλιών και Παλαιστινίων. Είναι λοιπόν συγκεχημένη κατάσταση και η κατάσταση αυτή αναφέρεται και ε, στα εμπορεύματα που μετέφερε αυτός ο στολίσκος που μπορούσαν να έχουν διέλθει ε, διαξηράς ε, για να αποφύγουν τον αποκλεισμό το να υπάρξει μία διεθνής έρευνα με ε, δύο τουλάχιστον διεθνείς εκπροσώπους δεν είναι κακό αλλά το Ισραήλ μεταξύ μας κύριε Πρόεδρε επιθυμεί να εξασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν πλέον επιθέσεις με ε, πυράβλους άπαξ και αρθεί ο αποκλεισμός. Κάνω λοιπόν μία έκκληση προς την ύπατη εκπρόσωπό μας για να σταματήσει η τρομοκρατία. Το η PLO να αναγνωρίσει ε, ε, το κράτος Ισραήλ και ε, να ελευθερώσει τον κρατούμενο. Κυρία Άστον, ε, είπατε κι εσείς ότι θα πρέπει να κάνετε προσπάθειες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμευτήκατε προς αυτό και εμείς ε, θα παρακολουθούμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι γίνεται και από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν, γιατί με την επίθεση του στο στολίσκο της ελευθερίας δεν είναι πλέον ατιμόρυτο το Ισραήλ όταν κάνει ουσιαστικά επίθεση κατά της νομιμότητας και στρέφεται κατά του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου. Το διεθνές ε, δίκαιο ε, καταπατείται ε, με αποτρόπαιο τρόπο προασπιζόμενο υποθέτω το Ισραήλ τα δικαιώματα και την ασφάλειά του. Έχουν θεσπιστεί, αυτοθεσπιστεί από το Ισραήλ ανώτατα όρια πάρα πολύ υψηλά και αυστηρά. Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά αυτά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα από το Συμβούλιο να γίνουν κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, διεθνή έρευνα, η οποία θα είναι αξιόπιστη ε, για την επίθεση αυτή, για το ρεσάλτο αυτό ουσιαστικά. Επίση, η άρση του αποκλεισμού και όχι μόνο αυτό το σύστημα των ε, καταλόγων και έπειτα διεθνή αναγνώριση ενό βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτου. Ο κύριος Μποντής για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, αυτή η επίθεση ε, προς τους πολίτες από τους Ισραηλούς, Ισραηλινούς στρατιωτικούς πρέπει να ερευνηθεί. Αλλά μπορούμε να, ε, να ε, έχουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή αυτή που εμπλέκεται, διότι η επίθεση έγινε σε διεθνή ύδατα ενδιαφέρει την διεθνή κοινότητα και την Ευρώπη, ιδίω στις παράκτιες χώρες της Μεσογείου. Η Ευρώπη πρέπει να υψώσει τη φωνή της περισσότερο και να εμπλακεί στη διερεύνηση μιας πολιτικής λύσης που θα βασίζεται σε δύο κράτη, εκ των οποίων το καθένα θα έχει ένα μέρος της Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα. Η Ευρώπη κάνει πολλές προσπάθειες για να αναπτύξει τα παλαιστινιακά εδάφη Δυστυχώς όμως απέχει πολύ από την πολιτική διαδικασία που πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία αυτού του Παλαιστινιακού κράτους. Η, οικονομική και δημοσιονομική καλή θέληση την οποία εκδηλώνουμε δεν αρκεί πρέπει να εκφράσουμε και μία πολιτική θέληση και να λάβουμε τον χρόνο να υψώσουμε τη φωνή μας για να μας ακούσουν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο σύντομο χρονικό διάστημα να επαναλάβω τα όσα μας είπαν εδώ έξω έξι επιβιώσατε στις επίθεσεις Όχι μόνο μας θύμισαν πως εννέα άνθρωποι θα ε, σκοτώθηκαν, επτά παραμένουν βαρύ κατάσταση και 55 τραυματίστηκαν συνδεσμαχία ΜΚΟ από 32 διαφορετικές χώρες με χριστιανούς, μουσουλμάνους, βουδιστές, άθεους. Το φορτίο ήταν τελείως ανθρωπιστικό, είχε, αποτελούνταν από μεμονωμένες δωρεές και ήταν δεσμευμένο στην ε, μία βία. Ορισμένοι από αυτούς λοιπόν δολοφονήθηκαν και τώρα και ο χαρακτήρας αυτού της αποστολής ε, τώρα αυτή τη στιγμή δολοφονείται. Μας είπαν πως είχαν ε, έξι σκάφη έτοιμα για ένα νέο στολίσκο για τον Ιούλιο και ότι θα στείλουν τα σκάφη ακόμα και αν δεχτούν νέε επιθέσεις. Δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν λέξεις, αλλά να προβούν σε δράσεις ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και πρόεδρε, λένε ότι μια χώρα που επιβεβαιώνει το νόμιμο της δικαίωμα σε αυτοάμυνα, δεν πρέπει να ε, καταδικάζει τους άλλους που αυτοαμύνονται και ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Νόμο. President. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε αμερόληπτη διεθνή έρευνα όπως το ζητάμε μετά από αυτό το τραγικό γεγονός θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε τον... Ε, φτάσουμε βιαστικά σε συμπεράσματα. Εγώ θα πρόσεχα σήμερα και πριν να ισχυριστώ ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είχε καμία σχέση, οποιαδήποτε σχέση με ακραίες οργανώσεις ή με πολιτικές συνιστώσεις. Είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της συζήτηση σήμερα ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια ισορροπημένη προσόγγιση. Ενώ θυμίζουμε στο Ισραήλ και το ζητούμε άμεσα να άρει τον αποκλεισμό, καλούμε και την Χαμάς που έχει πάρει την εξουσία με στρατιωτικό τρόπο και αναγνωριστεί και, και αρνείται να αναγνωρίσει την ύπαρξη του Ισραήλ και το δικαίωμά του στο να υπάρχει, να πάψει και τις εχθροπραξίες. Θα πρέπει να συνδέονται όλα αυτά αξιόπιστα. Ζητάμε από εσά, κυρία Άστον, να προβείτε στην πρωτοβουλία, να διασφαλίσετε την διεθνή παρακολούθηση των, της λωρίδας της Γάζας ώστε να ε, εντωμεταξύ εμείς να μετασχηματίσουμε τελείως την πολιτική μας στη Μέση Ανατολή. Grazie, ma colleghi, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που καταδίκασαν την επίθεση στον στόλο που κατευθυνόταν προς την Γάζα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα δυσανάλογων ενεργειών στις οποίες πρέπει το Ισραήλ. Αυτές οι ενέργειες κατέληξαν σε τραγωδία και έτσι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκε συμπεριλαμβανομένων αυτών που πάντοτε ε, αναζητούν τη μετριοπάθεια. Δεν λέμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να προστατέψει τους πολίτες, της, τους πολίτες του, όμως αυτή η στάση που κρατά, ότι δηλαδή βγαίνουν και σκοτώνουν όποιον θέλουν όποτε θέλουν, αυτή είναι μια στάση που δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Και ε, γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που επιμένουν για να γίνει μια έρευνα, μια έρευνα που θα αντικατοπτρίζει τα στοιχεία και τα γεγονότα όπως έγιναν και να εξασφαλίσει ότι το Ισραήλ θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η σύγκρουση μεταξύ ε, του ανθρωπιστικού στολίσκου και των ε, δυνάμεων του Ισραήλ επεδίνωσαν την κατάσταση στην περιοχή. Χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια και δεν μπορούμε παρά να συλληπιθούμε τις οικογένειες των θυμάτων. Θα έπρεπε Πρέπει η χώρα αυτή να είναι πιο ανοιχτή στην διεθνή συνεργασία και στα Ηνωμένα Έθνη. Χαιρετίζω το ότι ε, το Ισραήλ θα καταρτήσει μία επιτροπή ερεύνης αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρχει διεθνή σύσταση της επιτροπής αυτής για να είναι αξιόπιστη και αντικειμενική. Συγχρόνως να υπάρξει ένας μηχανισμός για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα και τέλος ε, κυρία Πρόεδρε πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιζητήσει μία λύση με δύο κράτη και κάνω έκκληση σε όλους τους ενδιαφερομένους να συγκρατηθούν και να μην υπάρξει χλιμάκωση της βίας στην περιοχή. Επίσης σε συνεργασία με την ε, Επιτροπή Έρευνας θα πρέπει να προχωρήσει για τη διαδικασία ε, κύριε Πρόεδρε, μου λέγει η Γραμματεία ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για το Catch the Eye. Ε, θα πάρουμε δηλαδή μόνο 6-7 άτομα και λυπάμαι για όσους δεν μπορέσουν. Η κυρία Αντρικένε. Θα είμαι επίση και πάρα πολύ αυστηρός με το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ λίγες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, η βία ακόμη και αν καταλήγει σε απώλεια ζώων πάντοτε θα πρέπει να καταδικάζεται και να καταπολεμάται. Βέβαια ακόμη δεν έχει καθοριστεί ποιο ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε βία στην περίπτωση ε, του Ρεσάλτο του Ισραηλινού στο, στο Λίσκο της Ελευθερίας. Δεύτερον, Συγχαίρω τη Ισραήλ για την απόφαση του να συμπεριλάβει στην διαδικασία έρευνας δύο ε, υψηλόβαθμους παρατηρητές οι οποίοι θα ε, διασφαλίζουν ε, την αμεροληψία και τη διαφάνεια της διαδικασίας. Είναι μια σοφή απόφαση κατά την άποψή μου. θα πρέπει το Ισραήλ να επανεξετάσει το ενδεχόμενο της άρσης του αποκλεισμού με τη βοήθεια ε, της διεθνούς ε, κοινότητας. Τι θα πει η διεθνής κοινότητα βέβαια άμα αρχίζουν ε, οι ρουκέτες πάλι να ε, στοχεύουν άμαχους Ισραηλινούς και η ε, παραστατική οργάνωση, οι οργάνωση Χαμάς να κάνουν ποτρόπες πράξεις. Ο κύριος Ιντάλγου. Έχει, έχουν δολοφονηθεί ήρωες ε, του αλτροισμού, της αξιοπρέπειας. Μιλάμε επίσης ε, για την ε, όλη αυτή η κατάσταση στα σύνορα του 1967. Σίγουρα πρέπει να γίνει έρευνα και πρέπει να καταδικαστούν πολλά πράγματα. Πέραν του ψηφίσματος που θα ψηφίσουμε θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ηθικό δικαστήριο το οποίο θα κρίνει ε, και θα δικάσει το βίαιο καθεστώς και κράτος του Ισραήλ. Όπως το δικαστήριο Ράσιλ για τα κλίματα πολέμου. Η κυρία Ρίς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ισραηλινή παρέμβαση στην, στο Στολίσκο ήταν μια καταστροφή, καταστροφή από όλες τις απόψεις ε, και από την ανθρώπινη πλευρά δεν το αρνούμεθα. Δεν αρνούμεθα επίσης ότι το, θα πρέπει να αρθεί ο αποκλεισμό ε, και αυτό είναι προφανές. Αυτή το ψήφισμα σε 17 σημεία μείον ένα, γιατί το κοινοβούλιο μας δέχτηκε να αναφέρθει το κύριο Τσαλίτ δεν περιλαμβάνει καμία αμφισβήτηση των κομμάτων των επιβατών της ειρήνης. Μόνο κατηγόριες ακούγονται, όλοι γνωρίζουμε και δεν είναι παραπληροφόρηση κύριε Χαουίτ, είναι γεγονότα. Όλοι είδαμε τις, στοιχείες, τις εικόνες όπου όλοι καλούσαν ε, στη τζιχάντ και βλέπουμε και την δημόσια τηλεόραση της Βαβαρίας που αποδεικνύει πως υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους ε, αντισημίτες Ισλαμιστές της Τουρκίας και τους ε, ε, επιβάτες της ειρήνης γιατί το ίμιση της αλήθειας δεν είναι αλήθεια. Μικρό, μικρό. Μικρόφωνο. Wait, wait. Herr Präsident, ich teile die Kritik am Vorgehen Israels, wie sie meine Kollegen Συμφωνώ με τις επικρίσεις που εκφράζονται για το Ισραήλ και τα όσα είπε και ο κύριος Σαλαφράγκα αλλά αν η Ευρώπη θέλει να έχει κάποιο ρόλο, να υπάρχει στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να μείνει και να παραμείνει εταίρος του Ισραήλ, ακόμα και αν το επικρίνει. Η κριτική είναι αποδεκτή, αλλά όχι το μίσος προς το Ισραήλ. Και ακούω διάφορες φωνές ότι, που δείχνουν πως δημιουργείται μίσος. Αν καταγράφουμε μόνο τα εγκλήματα του Ισραήλ εδώ, αλλά αγνοούμε τα εγκλήματα της Χαμάς, δεν νομίζω πως μπορεί να είναι αποδεκτό κάτι τέτοιο. Και αν απλώς κατηγορούμε το Ισραήλ για γενοκτονία, δεν νομίζω πως ούτε και αυτό είναι αποδεκτό. Και αν θέλουμε να πούμε ότι λόγω των όσων κάνουμε εδώ είναι δύσκολο να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη καν του Ισραήλ και αυτό είναι πάλι απαράδεκτο. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσέξουμε να μην μπούμε από μόνοι μας στη γωνία και υποβαθμίσουμε την... σε δικές μας τις ενέργειες. Τάνοκ, λυπούμε βαθύτατα για την απώλεια ζώνας του μελών του του Στολίσκου, αλλά και αυτή η κατηγορία κατά του Ισραήλ επίσης δεν με βρίσκει σύμφωνο. Έχει κάνει λάθη το Ισραήλ. Εγώ πάντως θα περιμένω την, ε, τα αποτελέσματα της έρευνας που θα ε, συμπεριλάβουν και έναν Καναδό και Βρετανό εμπειρογνώμονα. Οι κομάντος ε, πυροβολήθηκαν επίσης και μάλλον δέχτηκαν επίθεση και πυροβόλησαν βρισκόμενοι σε αυτοάμενα. Σε αυτοάμενα γιατί τώρα η τουρκική κυβέρνηση ουσιαστικά ε, συνεργάστηκε για την ε, αποστολή, για την ιοπομπή αυτή και γιατί ε, μπήκαν σε αυτή την περιοχή που ήξεραν ότι κατά αυτά θα υπάρξει αντιπαράθεση. Ξέρουμε ότι και η Χαμάς είναι μια απαγορευμένη παράνομη οργάνωση η οποία επίσης θέλει να προμηθευτεί όπλα. Δεν θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Κύριος Μαρινέσκου για ένα λεπτό. Eh, e- Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε προωθεί και προάγει την ανθρωπιστική βοήθεια σε κάθε περιοχή που βιώνει τέτοιε κρίσει και οι κρίσει ποτέ δεν θα πρέπει να έχουν ω αποτέλεσμα την επιδείνωση συνθηκών διαβίωση ε, του πληθυσμού. Ωστόσο, πρέπει ξεκάθαρα να αντιδρούμε όταν ανθρωπιστικέ δραστηριότητε ε, τελικά δυσφημίζονται και χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν ε, τρομοκρατικέ δραστηριότητε και λαθρεμπόριο όπλων σε εμπόλεμε περιοχέ. Είναι το Ισραήλ ένα σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλού τομεί και αυτή την εταιρική σχέση με το Ισραήλ θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε για να βρούμε επικοδομητικού τρόπου με του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στην περιοχή. Δεν θέλουμε να κατηγορούμε ούτε και να υπερασπιζόμαστε, απλά να βρούμε μια μακροπρόθεσμη λύση. για ένα λεπτό. Εγώ από ένα ανθρωπιστικό κόμμα προέρχομαι, γι' αυτό και θα υπερασπίζομαι πάντοτε ε, τον άνθρωπο και θα καταδικάζω τη βία. Τη βία και τη Χαμά μεταξύ άλλων. αναγνωρίζω ότι η περίπτωση με την Ιωπομπή ήταν ένα ακόμη παράδειγμα τη ε, δυσανάλογη βία που χρησιμοποιεί συστηματικώ ε, το Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού με την συγκατάθεση τη διεθνού κοινότητα. Περιβολικέ φορέ η διεθνή κοινότητα στρέφει άλλου οφθαλμού τη. Κυρία Άστον, ε, σα παρακαλώ να δείξετε σθένο για να αρθεί αυτός ο αποκλεισμός για να σταματήσει η προοδευτική κατοχή αυτών των ε, ιστορικών εδαφών, για να γκρεμιστεί αυτό το τείχος το οποίο είναι πονίδιστο και για να γίνει η ειρνευτική αυτή διαδικασία πραγματικότητα με τη δημιουργία δύο κρατών γειτονικών. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Ε, η Ευρώπη και εκπροσωπή τη με τον τρόπο αυτό θα έχουν και αυτοί το σεβασμό τη διεθνού κοινότητα. Ευχαριστώ. Ε, με ε, Η κυρία Όκεν για ένα λεπτό. Er η Ευρώπη είναι φίλη του Ισραήλ. Πάντοτε είμαστε φίλοι. Αλλά δεν έχουμε φερθεί έτσι. Έχουμε αφήσει το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και να καταστρέφει τη δική του φήμη ουσιαστικά και την ασφάλειά του και την ειρηνική συμβίωσή του με τους γειτονικού του λαούς. Αυτή τη φορά όμως το Κοινοβούλιο, θα έλεγα, με αρκετή μεγάλη πλειοψηφία έχει δράσει αποφασιστικά. Και θα έλεγα, κυρία Άστον, εσείς έχετε τα μέσα και έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πραγματικά κάτι ώστε να σταματήσει το Ισραήλ να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση που θα οδηγήσει τελικά και στο τέλος τη Παλαιστίνης αλλά και στο τέλος του Ισραήλ. Ελπίζω να καταφέρουμε να υπερβούμε όλες αυτές τις ασαφείς αόριστες διελώσεις που κουνάμε το δάχτυλό μας χωρίς να κάνουμε τίποτα όμως επί της ουσίας. Εσείς έχετε τα μέσα, θα χρησιμοποιήσετε, το ελπίζουμε. zutiefst bedauerlich, dass es offensichtlich είναι πραγματικά λυπηρό ότι χρειάστηκε αυτό το τραγικό γεγονός για να συνειδητοποιήσουμε τις ενέργειες του και τις πράξεις του Ισραήλ. Είναι ωστόσο παράξενο πως ξαφνικά η τουρκική κυβέρνηση φαίνεται να δείχνει φροντίδα και καλοσύνη προς αυτή την στολίσκο. Παρ' όλα αυτά απέναντι σε αυτόν τον απάνθρωπο αποκλεισμό είναι λογικό οι μετριοπαθείς να δυσκολεύονται και οι ε, εξτρεμιστές να το ευχαριστιούνται. Το Ισραήλ Πάντως, από, ε, ε, ε, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να υπάρξει μια διεθνής επιτροπή για τη Γάζα και συμφωνώ με τον πρόεδρο χρειάζεται θάρρος οι εκκλήσεις είναι ωραίες αλλά εάν δεν συνδυάζονται με κυρώσεις δεν μπορούν να ισχύσουν θα είναι η κυρία Ντουράντ και η κυρία Βεϊράκ κυρία Ντουράντ για ένα λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Άστον, επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα τελευταίο στοιχείο. Εκατομμύρια ε, πολιτών της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης απαιτούν από την Ευρώπη μία αντίδραση η οποία να είναι αντίστοιχη της, της δικιάς τους αρνήσεως και υπάρχουν πάρα πολλά θύματα τα οποία δεν δέχονται πλέον να καταπατάτε το διεθνές δίκαιο. Ορισμένα άτομα βρίσκονται εδώ στο θεωρεί πρόκειται για νέους δεσμευμένους για την πρόθεση της ειρήνης και γι' αυτό το ψήφισμα το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο πρέπει να εφαρμοστεί και να μην υπάρχει παστική ε, αντιμετώπιση των νέων της Ευρώπης διότι στο τέλος θα πιστέψουν οι νέοι αυτοί ότι μόνο οι ακραίες θέσεις πρόκειται να δικαιωθούν. Παρακαλώ λοιπόν ότι έγινε αυτή τη φορά να καταλάβουμε καταλήξει και σας ευχαριστώ. Κυρία Ντεβεϊράκ, για ένα λεπτό. Είναι εδώ. Είναι εδώ η βία επίθεση ή στο πλοίο Μαρμαρά πρέπει να καταδικαστεί ε, και ε, να καταδικαστεί διότι πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο τιμωρείται ο λαός του Ισραήλ από τις πράξεις του κράτους γιατί απομακρύνεται ο τελικός στόχος ε, για την περιοχή. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει σταματήσει την πολιτική της ε, ε, ε, επιδείξεως ισχύω, παρόλο που το πλοίο Μαρμαρά δημιουργεί αμφιβολίες ως προ τον πραγματικό του στόχο και εδώ αναφερόμαστε στην προετοιμασία αυτής της αποστολής και θα πρέπει η κυβέρνηση του Ισραήλ να δεχθεί μία ουσιαστική συμμετοχή διεθνή για να μπορέσει να υπερισχύσει η ειρήνη στην περιοχή. Ευχαριστώ. Για να κλείσετε την συζήτηση. Ε, um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο για μένα ακούγοντας τη συζήτηση είναι πολύ ξεκάθαρο είναι η έκκλησή μας ε, και η συμφωνία μας ε, για μια αξιόπιστη έρευνα οι Ορισμένοι συμβουλευτέ έχουν τι πληροφορίε του, διαφωνούν ω προ τι απόψει του. Ε, το σαφέ όμω είναι το εξή. Έχουμε εννέα νεκρού και έχουμε ε, οικογένειε ε, που θρυνούν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η έρευνα που θα γίνει να είναι αξιόπιστη, να μπορούμε να την πιστέψουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που είναι σαφές για μένα είναι ότι θέλετε να είμαστε σε επαφή με όλους τους σημαντικούς εταίρους που έχουμε για να αποφασίσουμε ποια θα είναι τα επόμενά μας βήματα. Και θέλω να σε επιβεβαιώσω ότι θα είμαι και ήμουν σε επαφή αυτή εξ αρχή με την Τουρκία. Μιλώ επίση και με το Ισραήλ και χθε μίλησα ε, με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον ε, Μαχμουνταμπά και με την Αίγυπτο έχω επαφέ θα έρθει στι ε, Βρυξέλλε να με δει την Παρασκευή, μάλιστα και ο Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών. Έχω μιλήσει με την Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα, την κυρία Κλίντον και γι' αυτό και για άλλα θέματα και με το κουαρτέτο και με τον απεσταλμένο του, τον ε, κύριο Μπλερ, με τον οποίο μιλώ σχεδόν κάθε δύο-τρει ώρε, γιατί έχει πηγαίνω έλθει τρει φορέ πηγαινοελθει ελθει τρει εβδομάδα στο Ισραήλ και στη διάσκεψη κορυφή με τη Ρωσία τα συζητήσαμε με τη Ρωσία αλλά και με τα 27 κράτη-μέλη έχω συζητήσει τα σχετικά ε, στο, τη Δευτέρα σε μια μακρά διαρκεία συνεδρία με τους Υπουργούς Εξωτερικών. Επομένως ε, υπάρχει αυτό ο διάλογο, ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε πώ θα προχωρήσουμε. Το τρίτο σημείο έχει να κάνει με τη σημασία τη πολιτική και με την αναγνώριση αυτού που προσπαθούσα να πω πριν. Ποιε είναι οι φιλοδοξίε ε, που έχουμε. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να δω είναι είναι ε, το Ισραήλ να ζει σε ειρήνη και ασφάλεια και βέβαια θέλω ο ε, Ισραηλινός στρατιώτης να απελευθερωθεί. Έχω ε, πρόσφατα συναντήσει τον πατέρα του εδώ στο Στρασβούργο. Πάντως έχοντας επισκεφθεί όπως και άλλοι βέβαια βουλευτές στη Γάζα ε, κατανοώ ότι η μελλοντική ασφάλεια της περιοχής εξαρτάται εν μέρη και από την ικανότητα, τη δυνατότητα των κατοίκων της Γάζας να ζουν ήρεμα. Να έχουν δηλαδή πλέον το δικαίωμα στο θαύμα, να μπορέσουν να ριζώσουν στην περιοχή, να ανθούν οικονομικά, ευημερούν, να μπορούν να ταξιδεύουν όπως οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος. 80% των κατοίκων τη γάζα βασίζεται σε τρόφιμα τα οποία παρέχει διεθνή κοινότητα και τα περισσότερα μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Πολλοί άνθρωποι δεν εργάζονται και Όποτε ε, έχω πάει εκεί, μιλώ με την κοινωνία των πολιτών, με ευρωπιστικές οργανώσεις, με την κοινωνία των πολιτών και συζητώ μαζί τους για τις ανάγκες τους, ποιες θα πρέπει να είναι ανάγκες τους και είμαι απολύτως βέβαια ότι η ασφάλεια της περιοχής, η ασφάλεια και του Ισραήλ εξαρτάται από το τι μπορεί να γίνει τώρα για να προχωρήσουμε. Επομένω, έχω επικεντρώσει στο δικό μου έργο, ελπίζω να συμφωνήσουν και οι βουλευτές ότι έτσι έπρεπε να κάνω, στο τι πρέπει να γίνει. Μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και Έχω ε, μιλήσει πολύ ε, και με το κουαρτέτο για να αλλάξουμε αυτό τον κατάλογο από τα 120 νομίζω αγαθά και εμπορεύματα απλά σε ένα κατάλογο απαγορευμένων αγαθών τα οποία δεν θα πρέπει να ε, περνούν στη Γάζα και ελπίζω να έχουμε πρόοδο σε αυτό ίσως ακόμη και σήμερα και νομίζω ότι αυτό θα έχει τεράστια σημασία αν λάβει κανείς υπόψη την τεράστια ποσότητα εμπορευμάτων που δεν μπορούν ε, να περάσουν. Ότι μπορούν ε, να περάσουν τα λουλούδια παραδείγματο χάρη, αλλά δεν μπορούν να περάσουν σοκολάτα, δεν μπορούν να περάσουν γλυκά, ε, μπορούν να περάσουν φρούτα, αλλά όχι ξηρή καρπή και ούτω καθεξής. Έχετε μελετήσει, φαντάζομαι, το χάρτη τη περιοχή, όπω και εγώ. Πρέπει να δούμε τα διάφορα σημεία διέλευση. Και χθε είχαμε μια αποστολή να υποστηρίξουμε για το άνοιγμα του σημείου διέλευση Ράφα, ε, που τώρα δεν είναι επιχειρησιακό, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιτόπου. Έχω μιλήσει με ανθρώπου. Αν δείτε το Council το κάνει, υπάρχουν δυνατότητε και για αυτά τα ε, σημεία διέλευση να μπορέσουν να ανοίξουν. Και όποιοι έχετε μελετήσει θα δείτε ποιο είναι το πιο εύθολο. Το κάνει για τα αγαθά, ενώ το άλλο όμω σημείο διέλευση θα μπορούσε ίσω να ανοίξει πρώτο. Αλλά και άλλα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε στο τραπέζι ορισμένα ζητήματα και για να παράσχουμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι δυνατότητε ε, να επηρεάσει τα πράγματα. Να ανοίξουν οι σταθμοί μεθοριακοί, ε, να μπορεί να γίνει προμήθεια των αγαθών προς τους Παλαιστινίους. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά βέβαια γίνονται και με την υποστήριξη των συνομιλιών του γερουσιαστού Μίτσελ. Εγώ ενθαρρύνω και παροτρύνω όλους όσους ενδιαφέρονται και εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες ε, να ε, κάνουν πραγματικές ε, συνομιλίες, να έχουν πραγματικές διαπραγματεύσεις, ουσιαστικές. Εγώ πραγματικά νιώθω και το λέω με ειλικρίνεια ότι είναι πολύ σημαντικό τώρα να γίνουν τα επόμενα βήματα. Και ενώ η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη σε αυτή την κατάσταση, θέλουμε να μετριάσουμε τα προβλήματα στην Γάζα και αυτό νομίζω ότι θα συμβάλλει σε αυτό που θέλετε όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή σε μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ειρήνη, ώστε να μπορέσει ο κόσμος ε, να ζήσει τη ζωή του σύμφωνα με τις ε, αρχές του, σύμφωνα με τις αξίες του και να μεγαλώσουν τα παιδιά όλων με ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος για την παράτωση αυτής της ε, συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Madam High Representative, are going to be here until ε, about 7 o'clock. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, θα είστε εδώ μέχρι τις 7 αν δεν κάνω λάθος. Αν χρειάζεστε δύο λεπτά, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Όχι, ωραία. Να πάμε άμεσα στην επόμενη συζήτηση. Ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες θα προεδρεύσει τώρα.